στο Κοινοβούλιο. Και θα το εξετάσουμε δεόντως αυτό το αίτημα ε, οι συνάδελφοί μου και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περατώθηκε η συζήτηση. Στην ημερήσια διάταξη τώρα έχουμε την έκθεση LifeFit που αφορά την ανάθεση κατεξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων για θέσπιση ορισμένων μέτρων σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λάιχφριντ, για τέσσερα λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αλλά θα μιλήσω γερμανικά γιατί δεν θα μπορέσω να εκφράσω κάτι λογικό στην Ιταλική γλώσσα. Θέλω όμως να επωφεληθώ της ευκαιρίας ε, στην αρχή της ομιλίας μου και στην ολοκλήρηση του ελέγχου αυτού του φακέλου να ευχαριστώ ότι, ευχαριστήσω ότι η έκθεση αυτή μπόρεσε να διεξαχθεί στην ε, Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου ε, χωρίς προβλήματα και ελπίζω ότι ίδια πορεία επιτυχίας θα ακολουθήσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ρωμέλεια και ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Γραμματείας της Επιτροπής και της Σοσιαλιστικής Πολιτικής Ομάδας που με στήριξαν ανα πάσα στιγμή και ιδίως τους ε, άμεσα προσκύμενους συναδέλφους μου ε, και πραγματικά είμαι ευγνώμων. Η ε, εμπορική πολιτική σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας έγινε ε, μια πολιτική στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα συναπόφασης και βλέπουμε τι ε, προσόντα προσδίδει αυτή η ιδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πολιτική πολιτική. Πρέπει όμως ε, να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο και η παλιά επιτροπολογία δεν μπορεί να συνεχίσει και τώρα σύμφωνα με το πρώτο κανόνα όμνιμπους και τον δεύτερο κανόνα όμνιμπους διότι στην ε, αρχή είχαμε αναφερθεί στις νομοθετικής πράξεις και στη δεύτερη, μου, στη δεύτερη όμνιμπους ε, 2 τη δικιά μου έκθεση δηλαδή με τις κατεξουσιοδότηση πράξη και ε, θα χρειαστούν διαπραγματεύσεις για γρήγορη ολοκλήρωση. Το Συμβούλιο όμως δεν κάνει τίποτα, δεν παρίσταται και συμπεριφέρεται σε αυτά τα τεχνικά θέματα όπως και γενικότερα. Δηλαδή ε, δεν χρειάζεται πλέον να μιλάμε για τον προϋπολογισμό ο οποίος είναι δύσκολος ε, για να καταλήξει αλλά ε, βλέπουμε ότι και σε άλλα θέματα δεν αντιδρά το Συμβούλιο και αν οι εθνικοί εγωισμοί ε, και οι κυβερνήσεις ακολουθήσουν αυτήν την πολιτική περαιτέρω ε, δεν θα καταλήξουμε πουθενά υπάρχει ε, μία οικονομική σφαγή θα επιστρέψουν όλοι στα εθνικά τους νομίσματα και για όλα αυτά οφείλεται το Συμβούλιο, ευθύνεται το Συμβούλιο που που θα έπρεπε εδώ να εργαστεί σοβαρά και να εγκαταλείψει τους εθνικισμούς. Πρέπει να κατανείμουμε το τι μπορεί να αναλάβει η ιδία της ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα πρέπει να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να βρούμε μία σωστή μέση οδό και βάσει της προτάσεώς μου ε, το Κοινοβούλιο απεφάσισε πρώτα στην Επιτροπή και ελπίζω και συνέχεια στην Ολομέλεια ότι έφτασε η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιορίσει τη δραστηριότητά της στις κατεξουσιοδότηση πράξη και αυτό να περιοριστεί σε μία πενταετία για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος. Κατά τα άλλα νομίζω ότι καταλήξαμε στο σωστό αποτέλεσμα ε, σχετικά με τις ε, ε, αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και τις τεχνικές διατυπώσεις. Ελπίζω ότι αυτή η νομοθεσία θα μπορέσει να προωθηθεί και στην Ολομέλεια για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δράση μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Σαμέτα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Πρώτα απ' όλα ζητάω συγγνώμη εκ μέρους του Επιτρόπου Ντεγκούχτ που διαπραγματεύεται σήμερα το πρωί με τους Καναδούς ομολόγους του όσον αφορά τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τον Καναδά. Η Επιτροπή είναι ευγνώμων προς ε, εσάς και προς τον εισηγητή, τον ε, πρόεδρο της ε, Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και τους άλλους ευρωβουλευτές που δούλεψαν πάνω στην πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει πολλές τροπολογίες. Οι περισσότερες από αυτές είναι τροπολογίες που μπορούμε να δεχτούμε. Ιδιαίτερα μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή στην περίοδο, την χρονική της κατ' εξουσιοδότηση πράξης στα πέντε χρόνια. Όμως ορισμένες τροπολογίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, γιατί ορισμένες αποκλίνουν από την αμοιβαία κατανόηση όσον αφορά την κατεξουσιοδότη, της κατεξουσιοδότηση πράξης. Αυτό έχει να κάνει, για παράδειγμα, με τροπολογίε οι οποίε επιβάλλουν συγκεκριμένε υποχρεώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη, όσον αφορά την προετοιμασία των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Άλλε τροπολογίε ε, πάλι ε, μιλούν για μια διαφορετική περίοδο. Εμεί δεν μπορούμε να τις δεχτούμε εκτός εάν η επέκταση στην περίοδο αιτιολογείται από ιδιαιτερότητε στον σχετικό κανονισμό. Οι τροπολογίε με τις οποίες διαφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τέτοιες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει πως τελικά θα έχουμε επικοδομητικό διάλογο ε, κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου και θα καταλήξουμε σε λύση. Ολοκληρώνω ε, επιμένοντα στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά όλου ιδιαίτερα το δικό σα έργο για αυτό το θέμα. Προσβλέπουμε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε συμφωνία κατά τον τριμερή διάλογο. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα δώσω τον λόγο τώρα στους αγορητές που μιλούν εκ μέρους των πολιτικών τους ομάδων. Δεν νομίζω ότι είναι στην αίθουσα συνάδελφος Κίστοτ Ρόουλ. Δίνω λοιπόν, έχετε το λόγο για τους σοσιαλιστές, κύριε Κούτας, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω την πρόταση κανονισμού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα όπου τροποποιούμε δέκα κανονισμούς όσον αφορά την κοινή εμπορική πολιτική σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα ήθελα να συγχαρώ τον Γιώργ Λάικφριντ, τον συνάδελφό μου, για τη δουλειά που έκανε για να συντάξει αυτή την έκθεση. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα, πάρα πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Είναι πασίγνωστο ότι όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι υπεύθυνα για την έγκριση νομοθεσία, θέσπιση νομοθεσία. Όμω για πρώτη φορά η συνθήκη τη συμπεριλαμβάνει αυτές τις πράξεις ε, κατεξουσοδότηση σύμφωνα το άρθρο 290, όπου το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να αναθέσουν ε, αρμοδιότητες κατεξουσοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λαμβάνονται πιο αποδοτικές αποφάσεις. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν το δικαίωμα να άρουν αυτή την εξουσοδότηση ή να καθορίσουν χρονικά όρια για την εξουσοδότηση. Σχετικά με αυτό, στην έκθεση αυτή, ε, προσπαθούμε να επιτρέψουμε στο Κοινοβούλιο πρόσβαση σε συνεδριάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεδριάσει εμπειρογνωμόνων για καλύτερη εφαρμογή των κατοξιδότη συμπράξεων όσον αφορά την κοινή εμπορική πολιτική. Ταυτόχρονα, συμφωνώ με τον περιορισμό της εξοδότησης κατεξοδότηση αρμοδιοτήτων για πέντε χρόνια όσον αφορά τις εξουσίες που δίνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται να έχει μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον εκτελεστικό κλάδο του Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ε, συνάδελφε Σαλβίνη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένα πράγμα είναι τεχνική, δηλαδή δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα επιλογή στην εμπορική πολιτική και αυτό είναι καλό. Άλλο πράγμα όμω είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή αυτό που φοβόμαστε εμεί σαν εκπρόσωποι τη Λέγα του Βορρά και εκπρόσωποι τη περιοχή του Βορρά, τη χώρα μα, είναι οι επιλογές οι εμπορικές, η σταδιακή μείωση ε, των απαιτήσεων, η, η επομείωση των ε, βιομηχανικών πολιτικών η επικράτηση των πολυεθνικών. Είναι καλό το Κοινοβούλιο δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει επιλογέ. Δεν θέλουμε να γίνουμε σκλάβοι όμω των επιλογών μια βιομηχανική και οικονομική πολιτική που είναι παλιά πολιτική του ΠΟΕ, που ευνοεί τι μεγάλε εξωτερικέ δυνάμει χωρί να προασπίζεται πουδενή του δικού μα παραγωγού. Δεν ξέρω να ξέρετε πόσε είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που κλείνουν αυτή την περίοδο στη Λομβαρδία, στο Βένετο, για λόγου λόγω συμφωνιών εμπορικών που δεν προστατεύουν καθόλου το προϊόν μα μπορείτε να φανταστείτε ότι μόνο με την έρευνα και την καινοτομία θα πάμε μακριά ενώ ε, θα, υπάρχει, θα μείνουμε έρημος όπως στις χώρες της Ανατολής όπου δεν υπάρχει κανένα εμπορικό κέντρο που να μην ανήκει στις μεγάλες πολυεθνικές ή στις Βόρειας Ευρώπης ή της Αμερικής Ασίας. Εμείς δίνουμε και στους σαν κοινοβούλιο εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη δυνατότητα να κάνει επιλογές για την εμπορική πολιτική με την ελπίδα ότι θα εξυγχρονίσει, θα αναθεωρήσει ε, ε, την τοποθέτησή του αφορά τον παραγωγικό ιστό που ε, εξαλείφεται. Ε, κύριε Σαρδίνη, δεχόσαστε μια γαλάζια κάρτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε συνάδελφοι. Ίσως παρανόησα, αλλά πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποσυρθεί και πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη τα οποία διαπραγματεύονται εις τον ΠΟΕ θα τα καταφέρουν εκεί καλύτερα. Διότι πρέπει να σας πω, παρόλο που στηρίζω τον ΠΟΕ, ότι ε, η ε, διαπραγματεύονται διαπραγματευτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι των μεμονωμένων κρατών και ε, δεν υπάρχει τίποτα σχετικά με τον ποέτο το οποίο ε, διαπραγματεύεται βάσει των κατεξουσιοδότης συμπράξεων και σε αυτό συμφωνεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με κάθε σεβασμό για τη δική σας δουλειά και την εργασία άλλων. Εγώ θα ήθελα να δείτε ποια είναι η παραγωγική πραγματικότητα της Βόρειας Ιταλίας και πόσες συμφωνίες που συνάπτονται μέσω του ΠΟΕ ε, είναι, έχουν θετικά ερευνητικά αποτελέσματα τις επιχειρήσεις μας. Ε, σε μισή ωρίτσα θα μιλήσουμε για τα φωτοβολταϊκά τόξα τα κινέζικα, τις φωτοβολταϊκές συστοιχίες. έχει σήμερα ε, ε, η Ευρώπη δεν μετράει πολύ, σχεδόν μηδέν. Δεν ξέρω αν με μόνο με τα κάτι μέλη θα μετούσα περισσότερα. Αλλά η εμπορική πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την έποψη για τι επιχειρήσει μα είναι καταστροφική. Η ελεύθερη αγορά απλώ δεν εξυπηρετεί κανέναν. Σα ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Το λόγο έχει ο κύριο Σόλτ για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Λάιχτφριτ το οποίο τα κατάφερε πολύ καλά και μπόρεσε να συσπυρώσει όλες τις πολιτικές ομάδες. Από προσωπική μου πείρα ξέρω ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει δεν είναι εύκολες διότι ε, σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει αλλεργία κατά του θέματος των εξουσιοδότηση πράξεων. Ε, Βεβαίω, ε, παρόλο που σε δημόσιες ομιλίες προωθούν τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, το Συμβούλιο αρνούνται να σαρμόσουν τις νομοθετικές διαδικασίες και να καταστήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισότιμο νομοθέτη. Πλέον όμως δεν είναι, πλέον όμως δεν είναι μόνοι το μόνο το Συμβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γύρω από το τραπέζι και πιστεύω ότι έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο στην επεξεργασία αυτών των φακέλων και σας στηρίζω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Συνάδελφε Κουίστοτ Ρόουαλτ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Η νομοθεσία Omnibus 2, πέραν της ε, Omnibus 1, ε, την οποία εγώ είχα διαπραγματευτεί σαν εισηγήτρια, μία αναβάθμιση ε, της νομοθεσίας σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και η κατεξουσιοδότηση πράξης πλέον θα εφαρμοστούν στο εμπορικό δίκαιο. Αυτές οι κατεξουσιοδότηση πράξεις είναι πολύ σημαντικές για να μπορεί ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να εφαρμόσει πλήρως τα δικαιώματά του και οι ε, συνάδελφοι των Ευρωβουλευτών θα μπορούν μεν να συμμετέχουν στη συνεδρία Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά αυτό δεν αρκεί πρέπει οι πολιτικοί να μπορούν να επέμβουν και θα πρέπει να είναι ε, εγκαίρως ενήμεροι για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις ελπίζω ότι να ολοκληρηθεί ε, σύντομα η συζήτηση στο Συμβούλιο για να ξεκινήσουν οι συμβιβαστικές συζητήσεις για την νομοθεσία Omnibus 2 η οποία ε, έχει συζητηθεί και πρέπει να τονίσουμε ότι οι δύο νομοθεσίες Omnibus 1 και 2 αποτελούν ένα πακέτο και γι' αυτό ευχαριστώ τον συνάδελφο Λίχτφριντ πρώτον διότι παρουσίασε σωστά την έκθεσή του εις ε, το Συμβούλιο στην Ολομέλεια διότι ε, χρειαζόμαστε την κύρωση από την Ολομέλεια το συζητήσαμε και μαζί και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ε, για τις δύο νομοθεσίες παράλληλα. Συμφωνώ πλήρως με την άποψη του σοσιαλδημοκράτη συναδέλφου σχετικά με τον ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΠΟΕ. Οι 27 συσπηρωμένοι είναι καλύτερα από 27 αυτά μεμονωμένοι και νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικά συμφέροντα που παίζονται εις ε, τον ΠΟΕ και εις τις διεθνείς εκπροσωπήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Σούστα, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερως τον εισηγητή, τον Γιώργ Λάικ Φρίντ για αυτό το έγγραφο. Είναι μια έκθεση σημαντική διότι καθορίζει καλύτερα τις διοργανικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου επί ενός θέματος βεστή ευαισθήτου που είδε διευρυμένες τις εξουσίες του Κοινοβουλίου με, στον τομέα της ε, εμπορικής πολιτικής που αφαιρέθηκε από τη συναπόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα πρόβλημα ουσίας και δεν συνδέεται με, τα, με που θα αλλάξουμε τη σημερινή έκθεση και που εντάσσονται σε νέα πειθαρχία, σε νέο πλαίσιο. Αλλά εξετάζεται εδώ η σχέση που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από αυτή την έποψη, ενώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από την έκθεση του Γιώργ, είμαι πολύ λίγο ικανοποιημένος από τα λόγια που εξέφρασε ο Επίτροπος σε αυτή την αίθουσα. Υπάρχει ακόμα μια υπερβολή τεχνική θετικής προσέγγιση όσον αφορά τι σχέσει Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, Κοινοβουλίου. Υπάρχει εμφανής προσπάθεια πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου προσπάθεια συνεχή μειώσεως του, των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάσταση προ-Λισαβόνα. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό που έχουμε καθορίσει χρονικό όριο όσον αφορά την εξουσδότηση. Είναι σημαντικό να ζητούμε μεγαλύτερη διευκρίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να αυξηθεί ο έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτού. Μόνο έτσι μπορούμε εμεί να, δώσουμε, να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που έθεσε και ο κύριος Σαλβίνη. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αποκλειστικά θέματα της εμπορικής πολιτικής. Θα πρέπει να ενισχυθεί η εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν συγκρίση με τα μεμονωμένα κάτι μέλη. Πρέπει να είμαστε όμως πιο ισχυροί και εντός του ΠΟΕ Δηλαδή να έχουμε επίγνωση ότι χωρίς μεγαλύτερη προσοχή στην πραγματική οικονομία δεν θα βγούμε από την κρίση στην οποία έχουμε πέσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο για τη διαδικασία προσέχης προσοχής του Προέδρου. Λοιπόν, ξαναδίνω το λόγο στον Επίτροπο Σεμέτα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Για άλλη μια φορά θέλω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δουλειά που έχει κάνει πάνω σε αυτό το θέμα. Και υπενθυμίζω ότι πολλές από τις τροπολογίες που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν να κάνουν με θέματα τα οποία καλύπτονται από τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, είναι απόλυτα δεσμευμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει τη συμφωνία πλαίσιο του 2010 ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα και πιστεύει ότι η συμφωνία αυτή είναι και το καλύτερο πλαίσιο για να καθυσχαστούν οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου και όχι αυτή εδώ η νομοθετική πράξη που συζητάμε σήμερα. Όπως και να έχει πάντως το πράγμα, σημείωσα τις παρατηρήσεις σας και θα φροντίσω να τις ε, δώσω και στον Επίτροπο Ντεγκούχτ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει σε συζητήσεις μαζί σας στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία. Σας διαβεβαιώ ότι αποτελεί προτεραιότητα αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής, ο κύριος Λίχθριτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η εμπορική πολιτική ε, αποδεικνύει κάτι σαφέστατα ότι ε, μπορεί να μην συμφωνούμε με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια της ΠΟΕ και εγώ πιστεύω ότι πολλά έπρεπε να λειτουργήσουν διαφορετικά αλλά ένα είναι σαφές ότι το σύνολο της κοινή μας δύναμης είναι πολύ μεγαλύτερη από την μεμονωμένη ισχύ του κράθε κράτους μέλους και όποιος αυτό δεν το καταλαβαίνει και δεν το αναγνωρίζει οδηγεί στον κρεμό χώρα του διότι θα, μόνη της η χώρα αυτή θα θαυτεί και φαίνεται από την, ε, ε, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα ε, λειτουργούν πολύ καλύτερα. Βλέπουμε ότι το Συμβούλιο απουσιάζει, δεν μας ακούει και ευθύνεται για πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θέλω επίσης να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι καλό να λέει ότι δεν δέχονται το ένα ή το άλλο, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κοινοβούλιο είναι νομοθέτης και αν εμείς αποφασίσουμε σήμερα θα πρόκειται για κάτι αποφασισμένο, για μία νομοθετική πράση και το Συμβούλιο μετά θα έχει όλο το χρόνο συμβιβαστικά κάπου να αποφασίσει αλλά παρόλα αυτά θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τούδε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Όλο Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο και θα ψηφίσουμε στις 12. Περνάμε στο επόμενο σημείο.